τον Ρόμπερτ Εύανς και άλλους 40 υπογράφοντες μια αντίθεση ε, γραπτός για τη συζήτηση της συγκεκριμένη. Σύμφωνα πάντα με αυτά τα οποία λέει το άρθρο 94 εγγράφεται για συζήτηση και ψηφοφορία η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος. Τελευταίο λοιπόν θέμα θα είναι σήμερα το βράδυ το συγκεκριμένο ψήφισμα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 15η απογευματινή σήμερα. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Εύανς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε, τη Δευτέρα το απόγευμα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την κατάσταση την ανθρωπιστική στη Σρι Λάνκα, η οποία χειροτερεύει σύμφωνα με το άρθρο 91 η κατάσταση στο Σρι είναι πραγματικά εξαιρετικά σοβαρή. Αλλά το τι συμβαίνει στον τομέα τον ανθρωπιστικό δεν είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στο σώμα γύρω από το θέμα αυτό. Και γι' αυτό το προτιμότερο θα ήταν να κάνουμε μια κανονική συζήτηση, η οποία δεν είναι σοβαρό να γίνει σε αυτή τη συνάντηση, αλλά στην επόμενη συνεδρίασή μας μετά από δέκα ημέρες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα στηρίξει την πρόταση και μια και είμαστε ένα σοβαρό κοινοβουλευτικό σώμα, παρακαλώ να υποστηρίξουν το ψήφισμα αυτό για την επόμενη ολομέλεια έτσι ώστε να φανούμε εισάξιοι, θα έλεγα, του μεγέθους του προβλήματος κατά κάποιο τρόπο στη Σουηλάνκα. Θα ζητήσω λοιπόν πάρα πολύ σύντομα τους υπέρ και τους κατά. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης Evans. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης αυτής. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής. Κοιτάξτε, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα από την ανάταση των χειρών. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία. Να, για να δω λίγο γιατί φαίνεται ότι ε, βιάστηκα λίγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κονμπεντίτ που ζήτησε το λόγο και θα συνεχίσουμε μετά αρκετά γρήγορα ελπίζω. Κύριε Κονμπεντίτ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, πρόεδρε, όταν κάποιος προτείνει κάτι υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος αντιπροτείνει κάτι πριν την ψηφοφορία. Να πω λοιπόν ότι η κατάσταση στο Σρι Λάνκα είναι απλά δραματική. 150.000 κάτοικοι της χώρας αυτής είναι αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, στην Τύρμα. Δεν πρέπει λοιπόν να αφαιρέσουμε από την ημερήσια διάταξη σήμερα το Σρι για να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας και την αλληλεγγύη μας με τους αποκλεισμένους πληθυσμούς. Ευχαριστώ κύριε Κονπεντήτ, ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Έχετε λοιπόν την πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας και την πρόταση διατήρησης της ψηφοφορίας. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής, και είναι κατά της αναβολής. Καλώς. Κατά λοιπόν γίνεται, ε, δεν γίνεται δεκτή η πρόταση. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της Γκέριγκερ Ντεόντεμπεργκ. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Έκθεση Γκέριγκερ Ντεόντεμπεργκ. Ψηφίζουμε.